συμπεριληφθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης. Και προχωρούμε στην ημερήσια διάταξη. Κυρίες και κύριοι, πριν υπησέλθω στα επιμέρους σημεία της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να κάνω μια διαδικαστική δήλωση, παρατήρηση, ούτως ώστε να εκφράσω και μια παράκληση σε σχέση με τη διαδικαστική αυτή παρατήρηση. Πρόκειται για την έκθεση Προμπάρτσικ για την Ενεργειακή Ένωση που είναι έκθεση πρωτοβουλίας. Επί της έκθεσης αυτής πρωτοβουλίας συνολικά δέχτηκα πάνω από 200 τροπολογίες, τροπολογίες, ε, προτάσεις για ε, τμηματική ε, ψηφοφορία ή χωριστή ψηφοφορία. Πάνω από 200 αιτήσει. Παρακάλεσα την ομάδα που υπέβαλε τις περισσότερες από αυτές τις προτάσεις να ξαναδεί το θέμα και να δει αν όντως χρειάζονται, διότι αλλιώς την πρόταση θα την είχα αναπέμψει και θα είχα παρακαλέσει την Επιτροπή να ασχοληθεί πάλι με τις ε, τροπολογίες. Ευτυχώς ε, η ομάδα απέσυρε πολλές από τις ε, προτάσεις της, τα αιτήματά της, ούτως ώστε τώρα έχουμε 59 τροπολογίες, αλλά 40 εξακολουθούν να ζητούν χωριστή και τμηματική ψηφοφορία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, την Τρίτη θα πρέπει να ψηφίζομαι επί 45 λεπτά περίπου επί της έκθεσης αυτής της πρωτοβουλίας. Ε, από μία ώρα και δέκα λεπτά μειώσαμε το χρόνο στα 45 λεπτά. Σε κάθε ολομέλεια ε, εσείς ε, ασκείται πολύ μεγάλη κριτική εις ό,τι αφορά τη διάρκεια των ψηφοφοριών. Και έχετε δίκιο βέβαια. Παρακαλώ όμως ακριβώς για αυτό το λόγο να το ξαναδείτε πολύ προσεκτικά το θέμα. Δηλαδή να ε, ελέγχετε αν όντω οι ονομαστικές ψηφοφορίες χρειάζονται, αν κάθε τμηματική ψηφοφορία χρειάζεται. Αν γίνει αυτό νομίζω ότι όλοι θα ελαφρύνουμε το έργο μας παρά την υπέρβαση των ελάχιστων ε, ορίων. Ε, τώρα ε, είχα σκεφτεί να στείλω την, επιτροπή, την έκθεση πίσω στην Επιτροπή. Αν μπορούμε όμως να το προτείνουμε, ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην επιβαρύνονται πάρα πολύ οι επιτροπές που θα πρέπει να αναλαμβάνουν πάλι να ξαναβλέπουν τις εκθέσεις. Τώρα, το πρόγραμμα αυτή τη βδομάδα δεν προβλέπει καμία τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Τούρμες. Μια παρατήρηση σε ό,τι αφορά τις πολλές τροπολογίες ε, για την Ενεργειακή Ένωση. Επί ώρες, ε, ε, οι πέντε ομάδες που δημιουργήσαμε προσπαθούσαν να βρουν συμβιβαστικές τροπολογίες και πραγματικά για 40-50 τροπολογίες υπήρχαν 60 αιτήσει για τμηματικές τροπολογίες. Ε, ε, χρειάζεται μια στρατηγική ε, γιατί πολλές φορές η πολιτική ομάδα που υποβάλλει όλες αυτές τις αιτήσει δράει εκβιαστικά και η λύση δεν μπορεί να είναι μόνο η αναπομπή στις επιτροπές. Κύριε Τούρμες, γνωρίζετε ότι δεν έχω ιδιαίτερες επαφές με την ομάδα αυτή την ΕΝΕΦ. Η, η τάση αυτή που αναφέρατε, ότι έχει η ομάδα αυτή, ε, υπάρχει και σε άλλες ομάδες. Δηλαδή παρατηρείται μια παρόμοια τάση. Δεν θέλω να ε, ε εξαντλήσουμε το θέμα τώρα, ούτε θέλω να υπερασπιστώ την ΙΕΝΕΦ. Πάντως Σημειώνω ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική, άλλωστε αυτό ήταν και ο σκοπό τη ανακοίνωση που σα έκανα, γιατί εκεί αποσκοπώ να σκεφτούμε να δουλέψουμε αποτελεσματικότερα. Ε, κυρία Κάπλη. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μιλήσω για τις προσωπικές στάσεις, ο καθένας φέρεται όπως θέλει. Εμείς πάντως έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις πολλές τροπολογίες, ε, μειώσαμε τις σημειωματικές, τις ε, χωριστές. Πράγματι τα 45 λεπτά είναι πολλά, θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε κι άλλο το χρόνο των τμηματικών και χωριστών ε, τροπολογιών και ευχαριστούμε για την κατανόηση κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, όχι από ό,τι βλέπω. Οπότε το πρόγραμμα εργασίας για τη βδομάδα αυτή εγκρίνεται και προχωρούμε στο πρώτο σημείο ε, την ε, συζήτηση επί της έκθεσης που αναφέραμε του κυρίου Γκρομπάρτσικ για την πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση και του κυρίου Έριξον για την προετοιμασία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για το 2020. Ο κύριος Στοζενόφσκι έχει